Good morning, everyone. If there are no objections, the draft agenda... Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε θα εγκρίνουμε το σχέδιο της ημέρας διάταξης χωρίς αλλαγές και τροποποίησεις. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα, μια από τα πλησιάζουμε το τέλος της ε, θητείας, η απογευματινή συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου επιβεβαιώνεται γιατί δεν ήταν σίγουροι και θα κάνουμε κάποιες έκτακτες συναντήσεις. Στρασβούργο, 10 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα, 7 με 10 και την 5η 13 Σεπτεμβρίου, 9 με 12. Ε, ε, θα έχουμε ψηφορίες και στις δύο συναντήσεις. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες. Δεν έχουμε εστονικά, αλλά τον και κελτικά. Ω συνήθως ηλεκτρονικά ε, μπορεί να βρείτε τα έγγραφα της συνεδρίασης. Έχουμε την εφαρμογή με την Πριν αρχίσουμε το πρώτο μας μέσα της διάταξης, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους διερμηνείς. Γιατί έχουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα για βάση. Οπότε παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας, τόσο να ακούσετε. τα μεταλείπει τους θερμινείς σα πληροφορούν ότι λόγω τη ε, εργατική διαφορά για τις νέες συνθήκε εργασία που έχουν επιβληθεί μόνο εμ, ε, δεν θα παρασχεθεί διερμηνία μετά την ώρα που προβλέπεται στην ε, συνεδρίαση. Άρα η συνεδρίαση θα τελειώσει, η διερμηνία θα τελειώσει μάλλον την ώρα που προβλέπεται η λήξη συνεδρίασης. Okay, thank you very much. Πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο θέμα υπαριθμών 4 της σημερινής διατάξεως και έχουμε τώρα την συζήτηση αυτού του σχεδίου ε, εκθέσεως για τον κανονισμό των ομαστικών ποσοτήτων για τη διάθεση αγορά της ε, Ένωσης Σουτσού με απόσταξη σε άνθρωπο που καταφερλώνεται στην ε, Ιαπωνία και η υποφαινόμενη είναι η να σας πω κάποια παρατηρήσεις και κατόπιν να λάβω το λόγο οι σκιώδες εισηγητές. Οπότε να σας εξηγήσω με λίγα λόγια τι ισχύει ε, και πώς κατέληξε αυτόν τον κανονισμό. Όπως θα ξέρετε υπάρχει μια συμφωνία με την Ιαπωνία που είναι η μεγαλύτερη εμπορική σχέση που έχει εμπορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι τώρα θα ανοίξουμε μια μεγάλη αγορά. Θα υπάρξουν πάρα πολλές ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές και έτσι θα καταργηθούν οι περισσότεροι δασμοί που είναι μεγάλο κόστος. Ένα εκατομμύριο της για τις εξαγωγικές μας ε, εταιρείες προς την Ιαπωνία. Θα ανοίξει επομένω η αγορά της ε, Ιαπωνία που σημαίνει 127 εκατομμύρια καταναλωτές και θα έχουμε επομένω ε, αυτές τις ε, εξαγωγές για 200 προστατευμένα προϊόντα μας που θα εξαχθούν. Ε, τα προϊόντα το οποία διέπονται από τις γεωγραφικές ενδείξεις επίσης θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για διάφορους άλλους κλάδους και θα μπορούν να συμμετάσχουν οι, οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε διαγωνισμούς στην Ιαπωνία και μόλις ε, την εγκρίνει ε, το Συμβούλιο Συμφωνία θα έρθει σε εμά και θα τεθεί σε, σε λειτουργία ε, θα καλύπτει η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη πριν το τέλος της ισχύου τωρινής εντολής της Επιτροπής του 19. Με αυτή την πρόταση θέλουμε να υπάρχει μια εξαίρεση από τους κανόνες για το μέγεθος των φιαλών για το σοτσού μονής απόσταξης που είναι ένα αλκοολούχο ποτό που εμφιαλώνεται και παράγεται στην Ιαπωνία παραδοσιακά πολίτες ε, φιάλες των 720 μιλιλίτερ και 1800 επίσης μιλιλίτερ και δεν ε, είναι ποσότητες αυτές που τώρα προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η εξαίρεση ούτω ώστε να καλυφθεί από την εμπορική συμφωνία μπορεί να γίνει μόνο με κανονισμό γιατί θα πρέπει να ισχύσει ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη όταν τεθεί σε ισχύ η εμπορική συμφωνία ε, με την Ιαπωνία θεωρώ ότι εάν εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις που ζήτηκαν στις διαπραγματεύσεις, ούτω ώστε να καταργηθούν οι περισσότεροι δασμοί, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και έτσι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι αγρότες αλλά και οι καταναλωτές να ωφεληθούν από αυτή την συμφωνία το συντομότερο. Και γι' αυτό θα πρέπει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής χωρίς προπολογίες και η ίδια διαδικασία έχει προταθεί να ισχύσει και στο Συμβούλιο στην ε, έκτακτη συνεδρίαση ε, της ε, ε, Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας της 11ης ε, έκτου και υπάρχει τώρα η καταληκτική μερομή της 13ης Ιουνίου που χωρίς να έχει υποβληθεί κάποια ένσταση ευσενικής αντιπροσωπείας εξέπνευσε ε, και τώρα να δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις ηγητές για να τοποθετηθούν. Κυρία Μελιόρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ καλά παρουσιάσατε. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με τις ονομαστικές ποσότητες και το μέγεθος των μπουκαλιών του ποτού αυτού το οποίο παράγεται σε άμβυγα. Τα παραδοσιακά ε, μπουκάλια εκεί είναι ε, μεγέθους 4 γκο, κάθε γκο είναι 180 μιλιλίτρο, το οποίο σημαίνει ότι τα μπουκάλια αυτά έχουν χωρητικότητα 720 ή αντίστοιχα 1800 ml. Εάν πρόκειται να εμφιαλώνονται ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό ε, για τα ινοπνευματόδη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό και Αντίστοιχα, να επιμείνουμε στην προστασία των γεωγραφικών ονομασιών ε, για ε, το ε, κρασί στην Ιαπωνέζικη αγορά. Το σιότσου είναι είναι ο πνευματόδης ποτό που παράγεται από ρύζι ή άλλα υλικά. Και θα χρειαστεί μία εξαίρεση στην Οδηγία 2007 κάθετος 45. Αυτή τη στιγμή ε, επανεξετάζουμε τον κανονισμό για τα υνοπνευματόδη και γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στο νέο κανονισμό. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, ε, συμφωνούμε με το Συμβούλιο και γι' αυτό θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα και εύκολα να εγκρίνουμε το θέμα αυτό και η τροποποίηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ε, ημέρα ε, θέσης ε, σε ισχύ της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία. Ευχαριστώ κύριε Σπίρκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία εισηγήτρια. Το ECR πιστεύει ότι η εξαίρεση για το Σιότσιου αποτελεί σημαντικό βήμα δεδομένης της ε, Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τη Ιαπωνία. Ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν προϊόντα και οι υπηρεσίες ε, συνολικά αξίας 58 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ ε, και πιστεύουμε ότι η Συμφωνία Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης θα εξαλείψει τα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ECR επικροτεί την δυνατότητα να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος εμπορίου και γι' αυτό θα χρειαστούν ε, κάποιες εξαιρέσεις όπως είναι η συγκεκριμένη περίπτωση το σιότσου. Οι φιάλες με ονομαστική αξία 720 ml ή 1800 ml αντίστοιχα δεν επιτρέπονται αυτή τη στιγμή. Με την εξαίρεση αυτή όμως μπορεί να πετύχουμε κάποιες παραχωρήσεις, ε, κάποιες εκχωρήσεις όσον αφορά ε, τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, και να αποφύγουμε τους δασμούς για τα κρασιά και τα υνοπνευματόδη μας. Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό το έγγραφο αυτό, είναι σημαντική η εξαίρεση αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των κρασιών και εινοπνευματοδών. Θα θέλαμε λοιπόν να στηρίξουμε την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιλουέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε το τελευταίο δωδεκάμινο, όπως και άλλοι συναδελφοί μου, έχω εργαστεί ως εσκιώδης εισηγήτρια πάνω στον κανονισμό ε, για τα εινοπνευματόδη και έχω ασχοληθεί με διάφορα εινοπνευματόδη. Αλλά όταν ε, κατέληξε στο γραφείο μου αυτό το θέμα του Σιότσου, έπρεπε καταρχάς να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Το Σιότσου ε, παρασκευάζεται στην, παραδοσιακά στην Ιαπωνία. Και ε, ένα από τα βασικά μας ε, θέματα στον κανονισμό ε, για την οπνευματόδη είναι η προστασία παραδοσιακών προϊόντων και γι' αυτό πιστεύω ότι πολύ σωστά θα παράσχουμε την εξαίρεση αυτή. Άλλωστε δεν νομίζω ότι ακριβώς πρόκειται για εξαίρεση. Έχουμε και στην Ευρώπη γεωγραφικές ενδείξεις και γι' αυτό θα ε, συστήσω στην πολιτική μου ομάδα να εγκρίνει την πρόταση αυτή χωρίς τροποποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Εάν όχι... Θα δώσω το λόγο στην κυρία Καμεσμορένου που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές της Επιτροπής σας ε, για την έκθεσή σας ε, και για το γεγονός ότι επικροτείτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι πολύ σωστά παρουσιάσατε το πλαίσιο καθώς και τον ε, στόχο της πρότασης. Και η ευρωβουλευτές της Επιτροπής σας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Το συνολικό πλαίσιο είναι η Συμφωνία Οικονομικής και Εταιρικής Σχέσης που όπως γνωρίζετε θα υπογραφεί στην διάσκεψη κορυφής αρχές Ιουλίου. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο και είναι ιδανικό ή εν πάρα πολύ ευνοϊκό για τον τομέα αυτόν, για το ευρωπαϊκό εμπόριο γενικά, αλλά ιδιαίτερα για τον ε, τομέα γεωργικών ε, προϊόντων και τροφίμων και ιδιαίτερα για τον ε, τομέα των ποτών. Ε, δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο τομέας αυτός από τη θέση σε ισχύ θα ωφεληθεί από Τρει σειρέ μέτρων. Καταρχάς, μείωση των δασμών. Ε, οι δασμοί στα κρασιά αυτή τη στιγμή είναι 50%, ενώ ε, θα είναι 7% ε, μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα έχουμε κέρδος δηλαδή. Επίσης, με την Ιαπωνία καταφέραμε να εγκρίνουμε τις εινολογικές πρακτικές του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ήδη ε, αναφέρθηκε, καταφέραμε η Ιαπωνία να αλλάξει την νομοθεσία της, ε, να δεχτεί τις, ε, τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις μας, εκ των οποίων έχουμε πάνω από 2.130 εκ των οποίων θα προστατεύονται στη Ιαπωνία. Έτσι διασφαλίζουμε την αποκλειστικότητα των ενδείξεων. Όλα αυτά λοιπόν όπως αναφέρατε αποτελούν ε, πολύ σημαντική χώριση από πλευράς της Ιαπωνίας. Στο πλαίσιο αυτό το σιότσου λοιπόν αποτελεί πολύ μικρή υποχώρηση σε σχέση με τα ωφέλη. Ε, δεν ε, ήθελα να το περιγράψω έτσι, αλλά η νομοθεσία μας έτσι διασφαλίζει περισσότερη διαφάνεια για τους ε, καταναλωτές μας. Και εδώ πέρα μιλάμε για εξαίρεση αποκλειστικά για το μέγεθος ε, της ε, φιάλης ενός παραδοσιακού προϊόντος. Το μέγεθος ε, του, της φιάλης αυτής ε, δεν ε, επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστη αυτή η παραχώρηση, την οποία θέλαμε να ενσωματώσουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Φυσικά το υποβάλλουμε στο Κοινοβούλιο για τη συγκατάθεσή του. θα θέλαμε όμως να είναι έτοιμη η νομοθεσία αυτή κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Και ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό ήταν με τροποποίηση του κανονισμού 110. Ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να χειριστούμε το θέμα αυτό από διοικητικής άποψης, αλλά να δείξουμε και την ε, καλή μας διάθεση απέναντι στην Ιαπωνία, διότι αυτό είναι θέμα ε, που τους ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό για την Ιαπωνία. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός στόχος αυτού του μέτρου. Αναφέρθηκε τι είναι το σιότσου. Ε, παράγεται από γλυκοπατάτες, ρύζι, ε, βρώμη ή ε, ε κρυθάρι, ή άλλα προϊόντα. Πρόκειται λοιπόν για πολύ ειδικευμένο προϊόν. και 500 λίτρα το χρόνο υπολογίζεται να εξάγονται το χρόνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για πολύ περιορισμένης κατανάλωση ε, και πολύ ειδικό προϊόν. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε την καλή μας διάθεση απέναντι στη Ιαπωνία κατά τη θέση σε ισχύ της ε, Συμφωνίας Οικονομικής και Εταιρικής ε, σχέση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση αυτή που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο συμφωνίας που θα υπογραφεί τον Ιούλιο. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Πήγαμε και στο Συμβούλιο ζητώντα την υποστήριξή σα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που στηρίζετε την πρόταση αυτή, διότι πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί πολύ καλή ε, ευκαιρία για την βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μα με τη Ιαπωνία σε όλου του τομεί, αλλά ιδιαίτερα ε, για τον γεωργικό τομέα. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ την Επιτροπή σα. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του και ελπίζουμε η πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθεί σύντομα και χωρί τροπολογίε για να παραδώσουμε στη Ιαπωνία αυτά που συμφωνήθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Um, uh, Σας ευχαριστώ. Η προθεσμία εκδόση τροπολογιών είναι στις 22 Ιουνίου στις 11 και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τα τέλη Ιουλίου. Επομένως, ε, ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα στην ημερησία διάταξη και περνάμε στο επόμενο. Um, λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 5, εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας και Περού. Εδώ εξετάζουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μελά. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 29 ε, Νοεμβρίου το 2017 η Επιτροπή Ίντα ζήτησε έγκριση να ε, να συντάξει μια χρωματότηση ακριβώ για την εφαρμογή τη συμφωνία, εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και του Περού ε, για πέντε χρόνια εφαρμόστηκε προσωρινά η συμφωνία και η σημερινή ε, έκθεση έχει ως στόχο να αξιολογήσει την εφαρμογή της συμφωνίας σε σχέση με το αν εφαρμόστηκε το σχέδιο δράσης ή βιώσιμη ανάπτυξη. Από ό,τι φαίνεται ότι κατόπιν της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης και ιδίω τη τελευταία έκθεση της 10 Οκτωβρίου 2017 και των παρατηρήσεων ε, της κοινωνίας ε, των πολιτών ε, ε, η τελευταία ήταν του Δεκεμβρίου του 2016. Αυτή η Σύμφωνη Ελεύθερων Συναλλαγών δεν ε, έχει σεβαστεί τις υποσχέσεις της. Ο οικονομικός αντίκτυπος ε, δεν έχει επιτρέψει την ανάπτυξη τομέων που αναμέναμε στο δευτερογενούς και το τριτογενούς τομέα στις χώρες των Άνδεων, καθώς υπήρχε περισσότερο των οικονομικών δραστηριοτήτων η δυναμική, είχε αρνητικές συνέπειες ε, μειώθηκε η τιμή των πρώτων υλών και ε, δεν υπήρξε βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας αυτών των χωρών. Η ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περού και Κολομβίας ε, εντείνει αυτό το φαινόμενο. Δείχνει ότι η συμφωνία οθεί προς μία ακόμη πιο ασύμετρη ανάπτυξη. Επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κολομβία και στο Περού μας δείχνει ότι στόχοι που εγγράφονται στο τίτλο 9 της συμφωνίας ε, δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή λόγω αστάθειας και έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων. Στην Κολομβία η συμφωνία με τις ε, ΦΑΡΚ που ανεστάλλει από τη νέα Προεδρία και της οποίας η εφαρμογή θα έχει σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στην ανακατανομή των γεών ε, και στην εντατική χρήση τους ουσιαστικά έχει συνέπεια σε σχέση ε, με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργικής ε, παραγωγής και το πώς χρησιμοποιείται η γη. Ε, η αστάθεια στη Βενεζουέλα έχει οδηγήσει σε μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Κολομβία και μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπινης εκμετάλλευσης και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Περού. Οι πολυάριθμες σειράξ, συγκρούσεις ε, πολλές φορές ε, κοινωνικές βίες ε, συγκρούσεις, η παράνομη εξορρεκτική δραστηριότητα, η αποψήλωση, η πολύ μικρή προστασία των εργαζομένων και των συνδικάτων. Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να μην υπάρχει φασαρία παρακαλώ. Λοιπόν, μας αφήνουν ε, να σκεφτούμε ότι η περιστολή της οικονομίας αυτής της χώρας και το άνοιγμα της ε, οικονομίας, της πολυεθνικές θα διευρύνουν αυτά τα φαινόμενα και θα εμποδίσουν την βιώσιμη και την ε, ανάπτυξη της χώρας αυτής. Και ξέρουμε βέβαια από το 2006 έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά στην κτηνοτροφία, όμως είναι δύσκολο να γίνει σεβαστό αυτό τώρα. Η έκθεση της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών ε, ενώσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, δεν έχουν επικυρώσει τη συμφωνία αυτή έτσι λοιπόν δεν γίνονται σεβαστοί οι στόχοι του τίτλου 9. Θεωρώντας λοιπόν ότι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις αρχικές ασυμμετρίες της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης, κατά την άποψή μου δεν ε, ωφελεί ούτε ε, αυτές τις χώρες των Άνδεων, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή της, κυρίως ως προς ε, την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και βιώσιμων στόχων και ζητούμε από το Συμβούλιο να εισαγάγει μια νέα, να δώσει μια νέα εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να γίνει αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα στραφώ στους σκιώδεις συζήτητες, ο κύριος Γκάμπος. Πάνω στην ώρα. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη γιατί μόλις ε, ήρθα και δεν μπόρεσα να ακούσω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι θα αρχίσει αργότερα η συζήτηση. Έχουμε εδώ μία, ε, μία έκθεση που αφορά την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Κολομβίας και Περού. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σχετικά. Καταρχήν, η ομάδα μου πάντοτε θέλει να διευρύνει τις ε, δυνατότητες των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Η ιστορία μας δείχνει ότι κάποιες ανοιχτές εμπορικές σχέσεις ε, μας έφεραν περισσότερη ανάπτυξη και ευημερία και σταθερότητα από ότι ο προστατευτισμός, ε, σενάρια του παρελθόντος που ουσιαστικά δεν προωθούν τη συνεργασία. Δεύτερον, η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας και Περού αποτελεί ε, ένα μύθο στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις δύο χώρες. Αυτή η συμφωνία μας βοηθά να δημιουργήσουμε περισσότερο εμπόριο μεταξύ των δύο μερών και αποτελεί ένα παράγοντα κλειδί για την αύξηση της απασχολησιμότητας ε, αλλά και της οικονομίας των δύο χωρών τη τη οικονομία. Πρέπει να Θυμόμαστε ότι προβλέπει έναν ασύμετρο ρυθμό απελευθέρωση του εμπορίου, καθώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει πλήρω συμφωνία ε, πριν το 2023, ενώ οι άλλε δύο χώρε τη Δυτική Αμερική πρέπει να το κάνουν πριν το 2030. Αυτή η διαφοροποίηση είχε ως στόχο να δώσει χρόνο στου ευαίσθητου ε, τομεί των χωρών εταίρων για να προσαρμοστούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Τέταρτον, Κατά τον ίδιο τρόπο, το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το εμπόριο είναι ένα κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας και τονίζει την δέσμευση των μερών στο να σεβαστούν και να εφαρμόσουν ε, τις θεμελιώδεις εργασιακές αρχές ε, και τις πολυμερείς συμφωνίες που αφορούν το περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα τα επίπεδα προστασίας που έχουν προβλεφθεί στην Εθνική Νομοθεσία. Για όλους αυτούς ε, τους λόγους ε, και άλλους που δεν θα αναφέρω τώρα γιατί πιέζει ο χρόνος, είναι απαραίτητο τα ευρωπαϊκή ε, όργανα, από τα ευρωπαϊκά όργανα και κυρίως από εδώ, από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μας να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας και Περού. Προς αυτή την κατεύθυνση ε, ζητώ συγγνώμη κύριε Συγητρία που δεν μπόρεσα να ακούσω την παρέμβασή σας. Εμείς ε, δεν ε, συμφωνούμε με τη γραμμή που ακολουθείτε στην έκθεσή σας και θα εργαστούμε έτσι ώστε το αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της Επιτροπής να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση. Όπως πάντα όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπούς, να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να σχολιάσουν την έκθεση αυτή. Αν δεν θέλει κανείς ε, το λόγο, ο κύριος Γιώργης από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας ε, εκθέσω την άποψη της Κομισιόν για το θέμα. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία αυτή από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογήσει την εμπορική συμφωνία, ακόμη και αν δεν έχει τεθεί πλήρω ισχύ. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε και εμεί από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, είτε φέτο ε, ή του χρόνου, και εμεί θα προβούμε σε μια ενδιάμεση αξιολόγηση τη συμφωνία αυτή. Να κάνουμε κάποια σύντομα σχόλια για τα σημεία που είναι υποσυζήτηση. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι για το αν πρόκειται για μια συμφωνία που έχει ωφελήσει την Κολομβία και το Περού να αναπτυχθούν προς μια πιο αηφόρη οικονομία και αν ε, τι έχει βοηθήσει στην οικονομική τους ανάπτυξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αν δούμε τα αποτελέσματα της συμφωνίας, είναι προφανές ότι η συμφωνία έχει βοηθήσει την Κολομβία και το Περού να απομακρυνθούν από μια οικονομία που βασιζόταν ε, ξεκαθαρά στις πρώτες ύλες προς μια οικονομία όπου υπάρχει προσθέμενη αξία, υπάρχει δυνατότητα για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις να συμμετέχουν και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αριθμητικά στοιχεία ως προς την αύξηση των ΜΜΕ στην Κολομβία και στο Περού που συμμετέχουν στις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης και διαφοροποίηση των εμπορικών ροών. Λιγότερες προτεσίλες λοιπόν και περισσότερα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα μετοποίηση από τις δύο χώρες. Το άλλο κύριο σημείο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με το δεύτερο σημείο στο σχέδιο έκθεσης που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και τα εργασιακά πρότυπα. Υπάρχουν ε, προκλήσεις ε, σε αυτές τις χώρες και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Με αυτή τη συμφωνία έχουμε δώσει σε αυτούς μας μια δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με αυτές τις χώρες και έχουμε δώσει και μια φωνή, ένα φόρουμ για την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές, ε, να υπάρχει με περισσότερος διάλογος, να μπουν σε περισσότερο διάλογο με τις κυβερνήσεις τους και σε διάλογο μαζί μας. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι νωρίτερα φέτος είχαμε έναν ε, συνασπισμό Περουβιανών ΜΚΟ που μας ε, παραπονέθηκαν σε σχέση με μη πλήρη, μη πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας από το Περού. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, όμως ε, από τη δική μας σκοπιά εμείς πέντε χρόνια μετά βλέπουμε ότι η συμφωνία δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις χώρες αυτές να έχουν πιο υφόρες οικονομίες και βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσει και τη δυνατότητά μας να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε και να οθήσουμε αυτές τις κυβερνήσεις προς ε, την κατεύθυνση μεγαλύτερου σεβασμού των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαλάν αν θέλετε να σχολιάσετε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Ναι, πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Με βάση τη θέση του κ. Καμπίου, κατάλαβα τι θέλουν και οι άλλε πολιτικέ ομάδε, αλλά κατάλαβα γιατί θέλω να πει η Επιτροπή και είναι σαφέ ότι πρόκειται να προσπαθήσουμε ε, επί τη βάση των τροπολογιών. Ε, πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, αυτό το θέμα, όπως ε, το έχει πει και η Ίντα και εμείς με τίποτα δεν είμαστε κατά των ελευθερών συναλλαγών με τις φίλες χώρες, ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να εισφέρουν, οπότε αυτές οι δημιουργίες μπορούν τις βοηθήσουν. Πάντω δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα σημάδια από τι διμερεί σχέσει, οπότε θα πρέπει να έχουμε και πίσω ρήτρε διαφύλαξη, κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο, λόγω ακριβώ των ε, σημερινών δυσκολιών και γι' αυτό περιμένω ανυπόμονα, περιμένω και με καλή διάθεση τις ε, τροπολογία και να συνεργαστούμε όλου του συναδέλφου. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους. Και σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η κυρία Βαλιάν. 3 Ιουλίου στις 11 η ώρα, εκπνέει η προθεσμία της ε, τροπολογίας, θα ψήμουν τον Οκτώβριο και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Στην Ίντα δεν θα ψηφιστεί τον Νοέμβριο. Και τώρα προχωρούμε. Έχουμε την ε, Κύριε Αντάλη εδώ. Για το επόμενο θέμα. Which is the post 2020 CO2 emission standards for new passenger cars and light commercial. Πρώτο επίδοση για τι εκπομπέ από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και σύντηση των τροπολογιών. Θα πρέπει να περιμένουμε την κυρία Ντάλη λίγα λεπτά. Πρέπει να σας ενημερώσω στο μεταξύ ότι χθε το βράδυ έκλεισε οι διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση στον τομέα της ε, ενέργειας. Με τον κύριο Ρούγκερ Μέτσκι Ε, που ενημερωνόμαστε για το τι έγινε. Να κύριε Αντάλη, λοιπόν, κύριε Αντάλη σας περιμένω τόσο ώστε να ξεκινήσει αυτή η ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις τροπολογίες όσον αφορά το θέμα. Thanks a lot. Um, Chair, thank you to the colleagues and thank you to the shadow rapporteur. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους σκιώδες εισηγητές που παρήσανται στην ε, συνάντησή μας, όπως ακριβώς και περίμεναμε. Αυτή η έκθεση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τώρα αυτές τις τροπολογίες. Περίπου 700 και επομένως τώρα βρισκόμαστε στην φάση της διαπραγμάτευσης για αυτές τις ε, τροπολογίες με τις πολιτικές ομάδες. Όπως θα περιμένει κανείς, περισσότερες τροπολογίες αφορούν τους ε, στόχους για το διοξίδιο και επίσης για τα αυτοκίνητα χαμηλών μηδενικών εκπομπών. Θέλουν ε, ε, μεγαλύτερου στόχου, υψηλότερου για το 25 και το 30. Πιο ψηλού από ό,τι πρότεινε Επιτροπή. Και έχουμε κάποιε τροπολογίε οι οποίε ζητούν για πιο αυστηρού στόχου για τα αυτοκίνητα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Για άλλε τροπολογίε λένε ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο μηχανισμό ε, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλοι ζητούν ένα σύστημα μπόνου μάλλον για αυτά τα θέματα και κοιτώντας τις ε, τροπολογίες προκύπτει σαφώς ότι η πρόθεση των συνέργων είναι στο να μην έχουμε παραθυράκια στο σύστημα ε, ιδίως όσον αφορά ε, την μετακίνηση του συστήματος το, των δοκιμών από NEDC προς το WLTP και σου λέμε με τις ε, εξαιρέσεις, τις παραμέτρους, ε, το πώς ε, σιγά σιγά θα καταργηθούν τα ρητά καύσιμα. Τέλος πάντων, όλα αυτά πρόκειται να συζητηθούν στις συναντήσεις με τους οικειοδησίγητες, οπότε θα μπορώ τώρα να σας πω ότι αυτό το οποίο θέλω είναι να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες για όλα τα μείζωνα θέματα του κανονισμού. Οπότε να σας τονίσω ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κανονισμού είναι αυτός ο υποχρεωτικός στόχος του 2025 και αν δεν υπάρξει ένας τέτοιος στόχος 35 γραμμάρια ανά που βλέπετε τώρα το 2021 θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 29. Οπότε, ε, αν δεν θεσπιστεί ο στόχο του 2025, αυτό είναι ένα κίνδυνο στο οποίο τρέχουμε. Γιατί συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα έχουμε το μισό του στόχου που θέλουμε. Οπότε αυτό δεν θα συνάδει σε αυτό το οποίο πριν από λίγου μήνε συμφωνήσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει να είναι πρώτο-πρώτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να γίνει η σχετική μελέτη για τι εκπομπέ. Αλλιώ τα κράτη-μέλη δεν θα είναι η θέση να μπορέσουν να τήρησουν του στόχου για το κλίμα. Είναι φανερό ότι έχουμε και κάποιε χώρε που κατάλαβαν τον κίνδυνο και είναι σε διαφορετικού βαθμού προετοιμασμένε και έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να τα καταφέρουμε για αυτή την νομοθεσία. Να σας πω τώρα για τους εργαζομένους. Χρειάζεται να προστατευτούν. Πιστεύω και ακόμη γι' αυτό θεωρείται νομοθεσία για το κλίμα. Αυτό είναι και νομοθέτημα το οποίο θα προστατεύσει τους εργαζομένους, θα εξασφαλιστεί ότι θα είναι καλυμμένοι από αυτή την αλλαγή που πρέπει να συμβεί. Γιατί έχουμε κάποια οχήματα μηδενικών εκπομπών που είναι πιο εύκολο να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και κάποια άλλα αυτοκίνητα όπω τα υβριδικά τα οποία είναι πιο δύσκολο να κατασκευαστούν και αυτό έχει σχέση με την απασχόληση. Επίση ε, προβλέπεται μέχρι το 2030 θα αυξηθεί η απασχόληση γιατί έχουμε κάποιους κινητήρες βενζίνη. περίπλοκοι και θα αυξηθεί η παραγωγή των υβριδικών οχήματων. Επίσης αυξήθηκε η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας λόγω της ε, μετάβασης προς ε, τις χαμηλές εκπομπές και αυτό έχει σχέση με την απασχόληση οπότε θα πρέπει για όλη αυτή τη διαδρομή να προστατευτούν οι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Τώρα αλλάζουν οι δυναμικές σε εθνικό επίπεδο και ενδείξεις λένε ότι έχουμε κάποιες χώρες που θέλουν ε, υψηλότερα πρότυπα για το διοξείδιο του άνθρακος, ψηλότερους στόχους για τις χαμηλές εκπομπές και πολλές από αυτές τις χώρες διαχειρίζονται την αλλαγή στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αλυσίδα προσφοράς σε σχέση με τις ελληνικές πολιτικές και έχουμε και κάποια κράτη τα οποίοι έχουν σε θέση, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, αλλά θα πρέπει να δούμε τι λέει το γερμανικό Υπουργείο. το 2030 θα έχει μισή, 50% και το 2025 επίση και το, ο λόγος για το 2025 για τις χαμηλές εκπομπές το 2025 θα είναι μια δοκιμασία για τους παραγωγούς ε, αυτοκινήτων και βλέπετε επομένω ότι κάτι κινείται στα κράτη-μέλη. Επομένως και ο Υπουργός, ε, η Υπουργός Περιβάλλοντος καταλαβαίνει ότι θα πρέπει η χώρα της να πετύχει το στόχο του 42% για το 2030. Οπότε περιμένω να ανταλλάξουμε απόψεις με τους σκιώδες και τους συναδέλφους. Ε, Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρος. Και τώρα και οδησυγητές. Πρώτα ο κύριος Γκίζε και... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια, η κυρία ε, Είπε ότι πρόκειται για μάλλον τεχνικό θέμα, αλλά τη στιγμή που έχουμε 700 τροπολογίες ε, βλέπουμε ότι μάλλον είναι και πολιτικό το θέμα υπόθηκε και πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν του 2017 ε, είναι ε, πολύ φιλόδοξη με στόχο 20% μείωση μέχρι το 2030 και διάμεσο στόχο μείωση 15% μέχρι το 2020. Ε, θέλουμε λοιπόν εδώ αύξηση της φιλοδοξίας ε, στο 75% θέλουμε διαγραφή της παραμέτρου χρηστικότητας που αντιστοιχεί στο βάρος ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε αντικειμενικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει πρόταση του ΕΛΚ για την προστασία του κλίματος, αλλά οι συνέπειες ε, για την βιομηχανία και για την απασχόληση δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το είπε αυτό η συγγήτρια και περιμένω να το δείξει αυτό. Έχουμε λοιπόν ε, τον στόχο του 25% για το 2020 με θα πρέπει όμως να εξετάσουμε ποιες είναι οι συνέπειες για την απασχόληση. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τεχνολογική ουδετερότητα και να μην έχουμε στόχους μείωσης που να μας οδηγήσουν στο να μπορούμε να τους πετύχουμε μόνο με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, διότι τότε δεν θα έχουμε ενεργειακή ουδετερότητα. Και τελικά καταλήγω να έχω περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Ε, το ηλεκτρισμός από πού προέρχεται, παράγεται με βιώσιμο τρόπο, ε, ποια θα είναι η υποδομή φόρτισης, ε, θα μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση και όταν βλέπω τις τιμές του κοβαλτίου για την παραγωγή μπαταριών, φοβάμαι ότι θα έχουμε προβλήματα στην αγορά. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι στην καινοτομία, στην οποία όμως ανήκουν και οι αναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε σοφή νομοθεσία, να προστατεύσουμε το κλίμα, να διασφαλίσουμε όμως και την ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας μας, ε, καθώς και τη διασφάλιση της απασχόλησης. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλές λύσει αν ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αλλιώ θα αποτύχουμε. Και πρέπει να πω ότι δεν βρίσκω πολύ σοβαρή την προσέγγιση της ε, συναδέρφου Ντάλι που ε, παραθέτει ε, μια γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας. Εγώ θα μπορούσα όμως να σας παραθέσω μελέτες άλλων γερμανικών υπουργείων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκίζε και ο κύριος Πρόκτορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ντάλη για όλη τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να εκπλήσει κάποιους ότι μπορώ να στηρίξω όλες ε, τις προτάσεις της όχι όμως στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ρεαλιστικό και δεν, είναι, δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις που είναι σημαντικές για την ομάδα του ECR μετά από τις πρόσφατες συζητήσεις που είχαμε στις ε, συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Ε, θα ήθελα να πω ότι καταρχάς οι εξαιρέσει ε, για την προηγούμενη περίοδο θα πρέπει να διατηρηθούν και κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο. Οι καινοτόμοι κατασκευαστές θα πρέπει να προστατευτούν και θα ήταν καταστροφικό να εγκαταλείψουμε τις εξαιρέσεις ε, αυτές αυτή τη στιγμή. Επίση, ε, όσον αφορά το να είναι οικονομικά προσβάσιμα τα οχήματα για του καταναλωτέ, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει αναδρομικά να τιμωρείται ο καταναλωτή μέσω τη νομοθεσία. Η βελτίωση των προτύπων των οχημάτων ε, θα πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα ε, με υπολογισμό του εθνικού τζίρου για τα οχήματα. Κατά μέσο όρο αγοράζονται νέα οχήματα κάθε 11 χρόνια στην Ευρώπη. Υπάρχουν σημαντικέ περιφερειακέ διαφορέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα παράδειγμα, ε, ο αριθμός αυτός είναι μάλλον ε, κάθε πέντε χρόνια. Επίσης, ε, πάντα χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα ώστε τα νέα οχήματα να εισχωρήσουν στην αγορά. Και τα πρότυπα για τα οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις σχετικές υποδομές οι οποίες είναι τραγικά ανεπαρκείς αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ενώ σε κάποιες περιφέρειες ε, τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ε, ρεαλιστική επιλογή, σε άλλες περιοχές δεν είναι. Για παράδειγμα, σε υπαίθριες περιοχές, διότι είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν αυτές οι μεγάλες εκτάσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατανόηση αυτού του προβλήματος. Επίσης, πολλά λέγονται για τους κατασκευαστές ε, οχημάτων. Μόλις τώρα ήρθα από την Επιτροπή Τραν, την Επιτροπή Μεταφορών και άκουσα πολλές απόψεις συναδέλφων, μερικοί εκ των οποίων βρίσκονται εδώ τώρα και άκουσα και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσαμε λοιπόν ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων ε, θα πρέπει να τα καταφέρουν καλύτερα, να ε, ξεκαθαρίσουν την κατάσταση ε, όσον αφορά τις εκπομπές του, των οχημάτων με ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν όχι πολλά χρόνια, το 1990, προωθούσε την πώληση ε, αυτοκινήτων δίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ήταν 14% ε, ε, το ποσοστό των διζελοκίνητων, ενώ πέρσι το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 52%. Γιατί συμβαίνει αυτό πολλοί από εμά γνωρίζουν και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ενέργειες των νομοθετών εδώ και στα κράτη-μέλη προώθησαν την πώληση και κατασκευή διζελοκίνητων οχημάτων. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει όταν οι καταναλωτές ε, είναι ε, επιφυλακτικοί και καχύποπτοι όχι μόνο απέναντι στους ε, Κατασκευαστέ των οχημάτων, αλλά και απέναντι στου νομοθέτες όταν προωθούν ε, καινοτόμε τεχνολογίες. Πάντως, όπως είπα, Πρόεδρε, συμφωνώ με τι απόψει ε, της κυρίας Ντάλι. Ε, αυτό που με απασχολεί είναι το κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η στόχη εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται μια ρήτρα αναθεώρησης καθοδόν ε, θα ήταν χρήσιμη για να δούμε πού βρίσκεται η τεχνολογία, εάν δηλαδή ακολουθεί τους ρυθμούς της φιλοδοξίας μας η τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριο Στόρβαλς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε πολύ καλές ε, συναντήσεις ε, υπό την προεδρία της κυρίας Ντάλη. Οι δικές μου τροπολογίες ε, στόχευαν σε τρία πράγματα. Καταρχάς να έχουμε ένα σημαντικό και ηχηρό μήνυμα για το μέλλον και για τους στόχους για το 2025, το 2030 και μετά από αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τις δοκιμές ε, σε υποπραγματικές συνθήκες οδήγησης ε, και τρίτον ε, να έχουμε και μία προσέγγιση του συνολικού κύκλου ζωής ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να υπολογίζουμε τις εκπομπές από, από όλα τα στάδια ζωής της τεχνολογίας. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Εάν δεν καταφέρουμε να πιέσουμε τους κατασκευαστές ε, οχημάτων να ανανεώσουν την τεχνολογία, τότε ε, κινδυνεύουμε να μας ε, ρίξει στο περιθώριο η Κίνα, το οποίο θα ήταν μεγάλη καταστροφή. Γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε τους κατασκευαστές όσο γίνεται. Όχι όμως μέχρι θανάτου, ε. πρέπει όμως κάπως να τους πρόξουμε. κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Υπάρχει μια τάση και φοβάμαι ότι η τάση αυτή ε, έχει να κάνει με το ιδεολογικό υπόβαθρο των θεμάτων αυτών. Φαίνεται σαν όλα να πρέπει να γίνουν με βάση τα ε, οχήματα μηδενικών εκπομπών. Πολύ ωραία ιδέα, αλλά Δεν είμαι βέβαιος αν θα καταφέρουμε να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση την βιομηχανία και μάλιστα τόσο γρήγορα. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο πόσο θέλουμε να τους πιέσουμε και πόσο αντέχουν. Ακούσατε τον συνάδελφο Γκίζεκε. Ε, η βιομηχανία φαίνεται να μην θέλει να δέχεται καμία πίεση. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να τα εξισορροπήσουμε όλα αυτά είναι να έχουμε μία σημαντική γενική μείωση διοξιδίου του άνθρακα. Με βάση υπολογισμούς του συνολικού κύκλου ζωής. Διότι έτσι θα έχουμε μια καλή προσέγγιση, ένα καλό πλαίσιο. Έχω ακόμα ένα μικρό πρόβλημα. Ε, δεν θέλω να ηθικολογήσω, αλλά εάν εισάγουμε σύστημα bonus μάλους, κινδυνεύουμε να ανοίξουμε την πόρτα για προσεγγίσεις ε, μη λειτουργικέ. πολύ ωραίε, αλλά μη λειτουργικές. Ε, θα πρέπει νομίζω να συζητήσουμε ε, περισσότερο ει βάθος αυτό το σύστημα bonus μάλους στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και να βρούμε μια καλή λύση στο πρόβλημα. Πάντως είμαι βέβαιος ότι το καλό πνεύμα που επικράτησε και κατά τις προηγούμενε συζητήσει θα μα οδηγήσει σε σοφή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Χάρμς. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ντάλη για τον τρόπο που διεύθυνε τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να πω στον κύριο Γκίζα και ότι δεν μπορώ να δεχτώ η μία πλευρά να αρχίσει να λέει ότι εγώ μιλώ με βάση τα γεγονότα, εμείς οι άλλοι δηλαδή τι κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό των γεγονότων και ποιος αποφασίζει τελικά τι είναι αλήθεια. Πάντως είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις. Για τη δική μου πολιτική ομάδα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο στόχος μείωσης για το 2030. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που ακούσαμε πριν υποβάλει η κυρία Ντάλη την έκθεσή της είπαν ότι αυτό είναι ο βασικός κόμβος, αυτό είναι το κομβικό σημείο όπου θα πρέπει να δούμε τι μείωση μπορούμε να πετύχουμε με βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες και με, τις συμβατικές, και με τους συμβατικούς κινητήρες και με εναλλακτικές μορφές κινητικότητας. Ε, με αυτή τη βάση θα πρέπει να επιλέξουμε τις καινοτομίες, τις φιλικές ε, προς το κλίμα ε, για την επόμενη δεκαετία. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα αυτό. Ε, εγώ και η δική μου πολιτική ομάδα εξετάσαμε προσεκτικά το θέμα διότι ε, αλλάζουμε με τροπολογία ε, αυτό που έχουν συστήσει οι επιρογνώμονες. Ο στόχος του Παρισιού ήταν να μην έχουμε αύξηση της ε, θερμοκρασίας του πλανήτη πάνω από δύο βαθμούς. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μείωση ε, εκπομπών τουλάχιστον 60% και βλέπω τον ε, κύριο Γκίζα και να κουνάει το κεφάλι του αρνητικά, αλλά αυτό είναι το γεγονός. Το πώς θα διαπραγματευτούμε τα θέματα αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Επαναλαμβάνω, εμένα με ενδιαφέρει να εκμεταλλευτούμε αυτό το κομβικό σημείο, ώστε ε, να μην μετανιώσουμε σε δύο χρόνια που θα διαπιστώσουμε ότι ε, ο τομέας αυτός δεν έχει συμβάλει στο μετριασμό του κλίματος ε, όσο θα έπρεπε. Όσον αφορά το ύψος του στόχου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει ενδιάμεσος στόχος και αναθεώρηση. σε τέσσερα 5 χρόνια πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ενδιάμεσο στόχο και αναθεώρηση και σε αυτό συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Όσον αφορά την ηλεκτροκινητικότητα, αυτός είναι ένας τομέας με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, διότι και εδώ ισχύει Ε, εάν ε, δεν ενεργήσουμε τώρα, ε, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν καταφέρουμε εμείς να κατευθύνουμε την καινοτομία στον τομέα των οχημάτων με την νομοθεσία μας, τότε ας μου πει κάποιος πώς αλλιώς θα γίνει αυτό. Και στη συζήτηση αυτή, κύριε Γκίζε, και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενώ εμείς μιλάμε για ηλεκτροκινητικότητα ε, και ε, ε, απώλεια θέσεων απασχόλησης, Στην αυτοκινητοβιομηχανία αναφέρεται συνεχώς η αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Οι μελέτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ε, λένε ότι οι σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης ε, στον, ε, στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα οφείλονται στην ηλεκτροκινητικότητα, θα οφείλονται στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση. Επίσης, ε, να πούμε ότι ενδιαφέρον βρήκα στην ε, τελευταία συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι τα κοινωνικά ωφέλη από τους πιο φιλόδοξους στόχους το κοινωνικό κόστος των υψηλότερων στόχων δεν θα είναι μεγαλύτερο. Μάλιστα το κοινωνικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο αν είναι πιο φιλοδοξοί στόχη και αυτό προκύπτει από μία μελέτη της E-Delft. Από οικονομολόγους, ε, από ε, μηχανικούς και από άλλους. Αυτά ακούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες. Έχουν ε, διεξαχθεί πολύ ομαλά οι διαπραγματεύσεις και είναι χρήσιμες οι συζητήσεις. Ε, και μάλιστα όχι μόνο στο πλαίσιο των ε, επιμέρους κρατών μελών, όπως ακούμε. Είμαι σκιώδης η και για την ε, οδηγία για την για τα οχήματα και τα δύο θέματα αυτά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Οι προτάσεις μου λοιπόν, οι τροπολογίες μου ε, σχετίζονται μεταξύ τους. Ήμουν λιγότερο φιλόδοξη αρχικά, ενώ τώρα είμαι περισσότερο. Είμαι η μόνη σκιώδη εισηγήτρια που προέρχεται από περιοχές όπου κατασκευάζονται συμβατικά οχήματα και όπου ε, όλοι οι άνθρωποι εξαρτώνται απολύτω από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, οι περιβαλλοντικές πτυχές, οι κοινωνικές, ε, οι πτυχές που σχετίζονται με την υγεία φυσικά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Αλλά δυτικές επιχειρήσεις έχουν τις εγκαταστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, ε, ετοιμάζονται ε, να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, αλλά στις δικές τους χώρες, ενώ στις δικές μας χώρες κατασκευάζονται τα συμβατικά οχήματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ομαλή μετάβαση. δεν θα λυθεί το πρόβλημα εάν απλά χάσουμε όλες τις θέσεις απασχόλησης της χώρες μας, ενώ οι χώρες όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις ε, αυτές ε, να εφαρμόζουν την καινοτομία. Και τελικά ε, ανατολικά της Γερμανίας μπορεί να έχουμε διζελοκίνητα οχήματα. Βλέπουμε αύξηση των ε, οχημάτων αυτών ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει να προσέξουμε, διότι αλλιώς δεν θα προστατεύσουμε ούτε την φύση, ούτε την υγεία των ανθρώπων. Θα ήθελα επίσης ε, ο στόχος του 2030 να είναι δεσμευτικός. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους ε, κατασκευαστές ε, οχημάτων εναλλακτικών ε, καυσίμων. Με ενδιαφέρει η τεχνολογική ουδετερότητα και γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογία σχετικά με τον συνολικό κύκλο ζωής όλων των οχημάτων. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τα εναλλακτικά καύσιμα και έχω υποβάλει επίσης μία τροπολογία για τις δοκιμές υποκανονικές συνθήκες οδήγησης. πέρα από ε, το διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να εξετάσουμε και τις ε, ε, εκπομπές οξυδίων του αζότου και οξυδίων του θείου. κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την υποστήριξη των καθαρών οχημάτων. Πιστεύω ότι δεν έχουμε πετύχει αρκετά κίνητρα για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει επαρκής υποδομή και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα αυτό. Βλέπουμε αύξηση των στόχων για τα κράτη-μέλη. Ε, προσβλέπω πάντως στην συνέχιση των συζητήσεων. Η έγκριση του εγγράφου αυτού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, στην κοινωνική πολιτική σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να το αγνοούμε αυτό και να μιλάμε μόνο για μείωση ε, των επομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είδαμε Άλλωστε ότι στηρίξαμε στο παρελθόν διζελοκίνητα οχήματα, ε, είδαμε ότι στηρίξαμε τα βιοκαύσιμα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που ήταν ανοιχτή απέναντι στις τροπολογίες μας ε, και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ισορροπημένο συμβιβασμό και να μην οπεφεληθούν μόνο κάποιες χώρες από ε, την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστούμε κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της μέχρι τώρα και για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουμε σήμερα επιτάπητους και για το πνεύμα συνεργασίας ε, που έχει δείξει. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα υποστηρίξουμε την γραμμή που έχει ακολουθήσει η εισηγητρία στην πρότασή της θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια βάσει και μέσα ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Θεωρώ βέβαια ότι ε, είναι κάπως ανησυχητικό ότι κάποιοι μοιοπικά ε, υποστηρίζουν ε, τα συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας που όλα αυτά τα έτη μας έχει δείξει ότι ήθελε να επιβραδύνει την εισαγωγή πιο αποτελεσματικών μέτρων μείωσης των εκπομπών και ε, τελικά δεν έχει κάνει και τίποτα για να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα που πραγματικά δεν θα ρηπαίνουν. Και επιτέλους ε, φτάνουμε σε αυτή την ιστορική στιγμή να εργαζόμαστε επί ενός σημαντικού κανονισμού που θα δώσει την ε, όθηση στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη ε, να ε, δράσει έτσι ώστε να μην χάσει και αυτό το ανταγωνιστικό προελέκτημα. Γιατί ξέρουμε ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου και ιδίως στην Κίνα η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία κάνει επενδύσεις για να γίνουν σεβαστοί κανόνες. Εγώ ως Ιταλίδα και Ευρωπαία θα ήθελα να μην χαθεί αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Να μην χαθεί ε, σε διαδικασίες απώλειας χρόνου. Θα πρέπει ε, να έχουμε ε, υψηλούς ε, στόχους ε, για το 2030 και επίσης είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε και τον ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών το 2025. Αυτό είναι πολύ σημαντική στιγμή για να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συμφωνώ με όσο είπε η και άλλοι συνάδελφοι για το θέμα της μετάβασης και επίση ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη μεταβατική φάση. Δεν ε, πρέπει να χάσουμε χρόνο. Θεωρώ ότι αν ε, δεν έχουμε η ε, υποχρεωτική διάταξη σε σχέση με την πώληση, όπως έχουμε προτείνει αυτή εμείς θα μπορούσε ε, να υπάρξει ένα σύστημα bonus μάλους, ένα διπλό σύστημα δηλαδή, ε, για να έχουμε ελάχιστους στόχους πώλησης αυτοκινήτων, ε, οχημάτων, μηδενικών εκπομπών. Έχουμε συζητήσει και το θέμα στους κοιόδης εισηγητές ο κύκλος ε, της ζωής ε, προκειμένου να υπάρχει ένα μια ξεκάθαρη εικόνα ε, σε όλο τον κύκλο της ζωής και της παραγωγής του οχήματος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα της εισαγωγής πραγματικών δοκιμών στο δρόμο. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό και για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όπως έχει γίνει και για άλλους ρήπους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα δύναμα σημεία του συστήματος ελέγχου, όμως ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους δρόμους ε, των πόλεων μας να έχουμε αυτοκίνητα που ρηπαίνουν περισσότερο από όσο λέγεται και η ρήπανση επιδεινώνεται σημαντικά στον χρόνο. Επομένως πρέπει να παρέμβουμε αποφασιστικά σε αυτό το θέμα, να έχουμε δοκιμές στο δρόμο και θα δούμε πώς ε, θα συζητήσουμε αυτό το θέμα περαιτέρω μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Και κλείνω ευχαριστώντας την εισηγήτρια. Ελπίζω ότι ο κανονισμός αυτός πράγματι θα μπορέσει να αποτελέσει μια καμπή για την Ευρώπη στον τομέα αυτό, γιατί το αξίζουν οι πολίτες που αγοράζουν ε, τα οχήματα, αλλά και οι πολίτες ε, που ζουν στις πόλεις, ε, γιατί είναι οι πιο ποινικοποιημένοι, γιατί έχουμε 400.000 θανάτους το χρόνο λόγω ατμοσφαιρικής ρήπανσης και δεν μπορούμε να γνωρούμε τον αριθμό αυτό. Εδώ ολοκληρώνουμε τις παρεμβάσεις από τους Κιώδης και θα προχωρήσουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους. Τρία άτομα έχουν ζητήσει το λόγο μέχρι τώρα. Παρακαλώ, αν θέλετε να σας φέρετε τη συζήτηση, κάτι ένα νεύμα. Ο κύριος Σαϊκούτ, καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον ε, και όπως ε, και συναδέλφους από το ΣΥΑΡ και εγώ ήμουν στην Επιτροπή Μεταφορών δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι ότι βλέπουμε μια τεράστια ορμή ε, Εντό στην Ευρώπη για την εφαρμογή τη συμφωνία των Παρισίων πρέπει να αυξήσουμε τι φιλοδοξίε, Ακόμη και χθε η Μέρκελ και Μακρόν είπαν ε, πολλά για διάφορα, αλλά είπαν και ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία τη μέχρι ε, την COP 2024. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι συζητούνται τα θέματα τη ενεργειακή αποδοτικότητα και των ενεργασίμων και φυσικά θα υπάρχουν και συνέπειε για το τι θα κάνουμε στον τομέα, για τον κανονισμό του επιμερισμού των ε, προσπαθειών και ε, φυσικά ένα τομέα είναι και οι μεταφορές και οι οδικές μεταφορές είναι κλειδί. Ξέρουμε ότι σε αυτόν τον κανονισμό τα μέτρα αποτελεσμα... τα πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα ως προς το κόστος θα πρέπει να ληφθούν στον τομέα των αυτοκινήτων. Τα αυτοκινήματα και οι εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα θεωρείται ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα ως προς το κόστος εκεί. Έτσι λοιπόν αν κάποιοι δεν θέλουν να κάνουμε τίποτα εκεί, τότε θα πρέπει να πληρώσουν, παραδείγματος χάρη το τίμημα, στη Γεωργία και προ προς συναδέλφους από το ΕΛΚ οι οποίοι τείνουν ε, να ισχυρίζονται ότι είναι συνεπείς. Αν θέλετε να είστε συνεπείς ε, και δεν θέλετε να πληρώσει το τίμημα η γεωργία, τότε θα πρέπει να είστε ε, σκληροί για την νομοθεσία για τα αυτοκίνητα, γιατί στέλνουμε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα στην αγορά γιατί πρέπει να κάνει μέχρι το 2030. Αν τα θαλασσώσουμε εδώ, τότε οι στόχοι επιμερισμού των προσπαθειών των χωρών θα αμφισβηθούν και τότε θα την πληρώσει η γεωργία. Μιλήστε με τους συναδέλφους από τη Γεωργία γιατί μετά θα ξυπνήσουμε, πολύ αργά όταν θα ξυπνήσουμε. Αυτά διακυβεύονται και θέλω να αναφερθώ και στον αγαπητό συνάδελφο Κίζεκε. Ε, είναι συναρπαστικό ότι τώρα σας ανησυχεί πάρα πολύ το ε, μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι καθαρό ή όχι. Είναι κρίμα που το ΕΛΚ δεν μας βοηθούσε να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές. Γιατί αν υπάρχει ε, συνεκτικότητα θα πρέπει φυσικά να καθαρίσεις και το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό θέλουμε πιο φιλόδοξους στόχους για τις ανανεώσιμες. Δυστυχώς εκεί έπρεπε να υποχωρήσουμε μέρει και λόγω του ΕΛΚ. Τώρα το ΕΛΚ μας λέει, α ναι, ε, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει πολύ λιγνίτης ε, στην ηλεκτρική ενέργεια και κάτι άλλο. Εκπληκτικό είναι ο ορισμό ε, τη ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο από τη ΣΥΑΡ ε, που ποτέ δεν ήταν ουδέτερο ω προ το θέμα τη τεχνολογία. Εμεί δίναμε κίνητρα στον δίζελ και ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε και τόσα κίνητρα του δίζελ γιατί γίνεται μέσω τη φορολογία και στη Γερμανία πάρα πολύ καιρό δίνονταν κίνητρα στον δίζελ Ισραήλ, όμως τώρα ο κύριος Γκίζεται ε, ουσιαστικά λέει, παραφράζοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνει πολύ φιλόδοξος ο στόχος, αν κάποιες χώρες δεν μπορούν να πετύχουν αυτό το στόχο. Ουάου, διευρύνεται ε, τώρα το θέμα της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας. Εγώ θα έλεγα ότι η μείωση του δεξιδιού του άνθρακα είναι ίδια για όλους, είναι ιδιαίτερα ουδέτερη για τεχνολογία και αν δεν μπορούν να τα καταφέρει τεχνολογία είναι πρόβλημα της τεχνολογίας. Τώρα όμως το αναστρέφεται. Αυτό δεν είναι τεχνολογική θέλετε πιο φιλόδοξο στόχο, γιατί φοβάστε ότι η βιομηχανία σας δίζελ δεν μπορεί να σεβαστεί το στόχο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αναστρέφετε τα επιχειρήματα. Πολύ απογοητευτικό, γιατί αν έχουμε μάθει κάτι από το Dieselgate, όπου ήσασταν συνσηγητής, είναι ότι ισχυροί στόχοι ε, ουσιαστικά προωθούν την καινοτομία στον τομέα και γι' αυτό πολλοί, γι αυτό πολλοί από την αυτοβιομηχανία λένε θέλουμε τώρα επενδύσεις εκτός Ευρώπης γιατί έχουμε μεγαλύτερη κανονιστική ε, ασφάλεια εκτός της Ευρώπης και ε, μιλάμε για τις δουλειές του μέλλοντος αν ε, δεν έχουμε κανονιστική ασφάλεια εντός της Ευρώπης τότε οι δουλειές θα είναι εκτός Ευρώπης αυτό διακυβεύεται εδώ γι' αυτό χρειαζόμαστε ξεκάθαρους φιλόδοξους στόχους για να έχουμε καλά αποτελέσματα για την απασχόληση και το κλίμα αν η τεχνολογία δεν μπορεί να τα καταφέρει και να του σεβαστεί τότε είναι πρόβλημα της τεχνολογίας Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να διακόψω κανέναν, αλλά προσπαθήστε, παρακαλώ, να περιοριστείτε, να περιοριστείτε το χρόνο, γιατί όπως ακούσατε θα είναι πολύ αυστηρή η διερμηνής ε, με το χρόνο σήμερα και έχουμε 15 λεπτά μόνο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Γκερμπράντι, ελπίζω να πήρατε το μήνυμα και ε, ποντάρω και το ότι είστε κουρασμένος από χθε το βράδυ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Γιατί είμαι κουρασμένος σημαίνει ότι θα μιλήσω πολύ αργά. Όχι, κάνω πλάκα. Σας ε, ευχαριστώ. Παίρνω σοβαρά τις παρατηρήσεις σας, όμως ε, δεν είμαι γνωστός ότι είμαι ακρηγορός στην Επιτροπή αυτή. Καταρχήν, μια παρατήρηση σας ε, απέναντι στο ΕΛΚ. Εγώ ε, εύχομαι να ήμασταν σε μια νέτη θέση για να μπορούσαμε να είμαστε χαλαροί για τους ε, στόχους ε, των εκπομπών διοξιδίου ανθρακά στα αυτοκίνητα. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ χαλαροί με αυτούς τους στόχους και πιστεύω ότι ο προηγούμενος ομιλητής ε, τα είπε καλά, δεν θα τα επαναλάβω. Λοιπόν, να τονίσω κάποια στοιχεία. Συχνά λέγεται ότι υπάρχει πολύ ε, αργή πρόσληψη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε του ε, ε, γεωταχή, αλλά σκεφτείτε, παραδείγματο χάρη, ε, τις δημόσιες αρχές, αυτές που έχουν ε, μεγάλου στόλου αυτοκινήτων, ε, που θέλουν να έχουν πιο καθαρού ε, στόλου αυτοκινήτων. Υπάρχει τεράστια ζήτηση και μάλιστα παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει επαρκή προσφορά. Περιμένουν για χρόνια ε, για να υπάρξει παροχή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπάρχει τεράστια ζήτηση λοιπόν. Ε, η ε, προσφορά είναι που δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Ένα άλλο επιχείρημα που είπε ο Μπάς είναι ότι ο κανονισμός σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετά αυστηρούς στόχους δεξιού του ανθρακά για πολλούς ε, όχι όμω για του τομεί ε, εμπορία εκπομπών. Και όπως ε, είπα ο κ. Κίζικ, θα πρέπει να ακούσουμε μόνο δεν θα πρέπει να ακούσουμε μόνο ε, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και τον Υπουργό Γεωργίας και τον Υπουργό Οικονομικών. Ξέρουν ότι αν δεν θέσουν στόχο στα αυτοκίνητα, ε, τότε θα υπάρχουν άλλοι τομεί που θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά για τη μείωση των εκπομπών. Αυτό σημαίνει το δομημένο περιβάλλον και ιδίω η γεωργία. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο παζάρι εδώ. Και δύο στοιχεία που θέλω να θέσω, γιατί έχω καταθέσει τροπολογίες γι' αυτά. Καταρχήν, να μετακινηθούμε ε, γρήγορα προς ε, τις δοκιμές R&D. Ε, να μην κάνουμε τις, τα ίδια λάθη ας έχουμε τις δοκιμές R&D το στομότερο δυνατό και το ίδιο ισχύει για ε, μία απαγόρευση ρητή ε, για τις ε, συσκευές για τις συσκευές που αλλοιώνουν τις εκπομπές. Αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη απαγόρευση και κατά τα λοιπά υποστηρίζω την εισηγήτρια και τους περισσότερους ομιλητές που άκουσα. Σας ευχαριστώ κύριο Σελίζε. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Μίρια Μτάλη για το σχέδιο έκθεσης. Και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους για την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στα γιοταχή οχήματα και τα ελαφρά ε, ε, επαγγελματικά οχήματα. Αλλά ε, τους στόχους εδώ μπροστά μας τους βρίσκω υπερβολικά φιλόδοξους και ελπίζω εδώ στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε ρεαλιστικούς στόχους. Ο Γιένς Γκίζε και εξέφρασε την θέση που έχει αποκρισταλωθεί εντός του ΕΛΚ. Ελπίζω λοιπόν από κοινού να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η κυρία Νταλή στην, ε, στο σχέδιο έκθεσή της ε, διαγράφει χωρίς να, τον χωρίς να την αντικαταστήσει την παράμετρο χρηστικότητας που αντιστοιχεί στο βάρος. Ε, έχουμε συζητήσει επί πολλά χρόνια το θέμα αυτό ε, στο πλαίσιο διαφόρων νομοθετημάτων. Είχαμε λοιπόν ένα συμβιβασμό, διότι ένα ε, όχημα με διπλάσιο βάρος δεν έχει και τις διπλάσιες εκπομπές. Υπάρχει εδώ μια βαλιστική καμπύλη και ίσως να μην είναι κατάλληλη η παράμετρος αυτή, μπορεί να χρησιμοποιήσει όμως κανείς άλλες παραμέτρους. Διότι, για παράδειγμα, ένα όχημα για έξι επιβάτες που χωράει μια ολόκληρη οικογένεια δεν θα πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις με ένα μικρό smart που χωράει μόνο ε, τον οδηγό λίγο πολύ. Ε, διαγραφή λοιπόν της παραμέτρου αυτής ε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε. Αποτελεί κόκκινη γραμμή αυτό για το ΕΛΚ. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Το άλλο θέμα είναι ο διάμεσο στόχος του 2020. Αν κατάλαβα καλά, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό ε, για την ε, τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού από ότι ο στόχος του 2003 το 2030 θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ε, όχι μόνο των νέων οχημάτων ε, αλλά και των παλαιών, του συνολικού στόλου. Ε, γι' αυτό μέχρι το 2030 θα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια προγραμματισμού λόγω των κύκλων δοκιμών και γι' αυτό οι κατασκευαστές δεν γνωρίζουν τι πρέπει να πετύχουν μέχρι το 2020. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς νομίζει ότι θα λειτουργήσει αυτό. Η κατεύθυνση είναι σαφής και γι' αυτό καταλαβαίνω και αυτό που είπε ο Νίλ Στόρβαλς. Ε, ίσως ε, θα πρέπει να έχουμε και στόχους για μετά το 2030, ώστε να μην προβάλλεται πάντα το επιχείρημα της ε, ασφάλειας προγραμματισμού. Η ερώτησή μου όμως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι... ότι ε, το να αναφερόμαστε στον κάθε κατασκευαστή είναι πολύ ε, σκληρό μέτρο. Ε, η αλλαγή του κύκλου δοκιμών μπορεί να συνεπάγεται υψηλές φιλοδοξίες για έναν κατασκευαστή και λιγότερες για άλλον ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα μπορούσαμε να βρούμε συμβιβασμό στο θέμα αυτό ώστε να μην έχουμε το δίλημα ότι αφενός ε, βραχυπρόθεσμα θα γνωρίζουμε ε, τι πρέπει να γίνει, ενώ από την άλλη να πρέπει να τηρήσουμε και τον ενδιάμεσο στόχο του 2025. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πρώτα-πρώτα να πω στους πράσινους φίλους ότι αυτή η φυκολογία μας ε, έχει αγανακτήσει αν έχουμε όλα αυτά τα δίζελ σήμερα. Ε, τόσα δίζελ είναι γιατί το ζητούσαν οι πράσινοι και ότι δεν θα έφερνε ε, το περισσότερο διοξίδιο και θα ήταν κλιματική λύση. ε, τελικά, ε, τι αυτό, κάποιος λέει ότι ξέρει την αλήθεια και αυτό μπορεί να ε, αλλάξει ανάλογα με την υποστημονική τεκμηρίωση που υπάρχει. Εντάξει, έχουμε τις προτάσεις το 25-30 της Κομισιόν, υπάρχει κάποια αισιοδοξία και φιλοδοξία σε αυτά και έτσι θα πρέπει αυτά να τα τηρήσουν οι αυτοκινητοβιομήχανοι και ότι εμείς επίσης θα πρέπει να κάνουμε κάποια προσπάθεια ούτως ώστε να έχουμε μείωση των εκπομπών. Αλλά ε, να φτάνουμε στο 70-75% με το 2030 ως μείωση, ε, αυτό είναι όνειρο απατηλό. Οπότε θα πρέπει έχουμε κάποιους στόχους που να μπορούμε να πετύχουμε. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος που αλλάζουμε τον ε, μηχανισμό του μπόνους για τα καθαρά αυτοκίνητα, αυτό το σύστημα που υπάρχει μπόνους μάλλον. Έτσι θα χαθεί η ουσία αυτού του μέτρου που είναι κίνητρο και όχι τιμωρία. Οπότε στο έχουμε στο κείμενο αυτό και άλλα τιμωρητικά στοιχεία. Το ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό μάλλον αυτοκίνητο τι είναι. Είναι η λύση, όχι κατά τα ΜΜΕ. Αλλά εδώ πέρα λένε εδώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι μόνο ηλεκτρικά και όχι άλλη τεχνολογία ως λύση. Άρα ας βρούμε κάποια λύση που να είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστούμε. Λέει πρώτος, οπότε τώρα τελείωσε ο κατάλογος των αγορητών. Ζητεί άλλο το λόγο. Και ο Ζούγκευ τώρα. Από την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Οπότε δεν θα επαναλάβω τα αυτά που λέει η πρότασή μας, μια που τα ξέρετε. Θεωρούμε ότι είναι φιλόδοξη και ότι είναι ισορροπημένη και ακούγοντας την συζήτηση σαφώς προκύπτει ότι όλοι στο ίδιο μήκο κύματο, να υπάρχει δηλαδή μια αυτοκινητοβιομηχανία ανταγωνιστική, να είναι καινοτόμα, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης εκεί να μην έχουμε εγκαταστάσει αλλού και επομένως πολλά από αυτά που θα πρέπει να επιλύσουμε είναι ε, θέματα τα οποία επιβάλλουν να προσαρμοστούμε στις ε, επερχόμενες ε, αλλαγές μέχρι το 2030. Οπότε και εμείς πολύ προσεκτικά εξετάζουμε όλες αυτές τις παραμέτρους για τους στόχους. Δεν τα είπαμε όλα στην μελέτη των επιπτώσεων, αλλά θα γίνει αυτό τώρα και έτσι θα γίνει κατανοητό ποιε θα είναι οι συνέπειε για του καταναλωτέ από πλευρά κόστου, ποιε είναι οι συνέπειε από πλευρά απασχόληση, ιδίω στην αυτοκινητοβιομηχανία και επίση ποιε είναι οι επιπτώσει όσον αφορά την ζήτηση σε άλλες, για άλλε τεχνολογίε Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει παραγωγή στην Ευρώπη. Θα πάρει αυτό κάποιο χρόνο. Κάποιες εταιρείες πάντως ευτυχώς έχουν πει ότι θέλουν να επενδύσουν σε αυτές τις τεχνολογίες. Αλλά βέβαια θα πρέπει αυτό να γίνει με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που θέλουμε να υπάρξει για τις μηδενικές εκπομπές. Να δούμε τι γίνεται με την υποδομή για τα αναλυτικά κάψιμα. Απαιτείται αυτή. Εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα, ιδίω στην Ήπεθρο. Αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Προσπαθήσαμε να τα λάβουμε υπόψη, προσπαθήσαμε έτσι να εκπονήσουμε την γνωστή πρόταση. Κάτι άλλο. Πώς θα γίνει η εφαρμογή. Όλα αυτά έχουν σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία, την ε, μετακίνηση προς τον WLTP, τη μέτρηση σε πραγματικές ε, συνθήκες, την ανάλυση του κύκλου ζωής και κάποιος είπε, νομίζω, ότι δεν θα πρέπει να είναι μια ζαριά αυτό, εκεί και ως έτυχε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα και με την ανάπτυξη του τεστ WLTP, και αυτό και αυτό μας πήρε 5 με 8 χρόνια για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Όχι, δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά κατα, καταφέρουμε να πάμε στο αντί. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Ένα σωρό δεδομένα, πρόσβαση στα δεδομένα. Θέματα ε, προστασία ιδιωτικού βίου, να βρούμε τα δεδομένα από όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Τι σημαίνουν αυτά τα δεδομένα. Α, και τα δεδομένα τι σημαίνει. Κάποιοι οδηγάνε γρήγορα και κάποιοι οδηγάνε πιο αργά. Να, πώς ε, μεταβάλλεται η κατανάλωση. Όμως, πώς αυτά όλα να τα αναγάγουμε στο τι κάνει ο κατασκευαστής. Επομένως θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο αυτό το πλαίσιο, αλλά χωρίς βιασύνη. Το 2024 θα γίνει μια αξιολόγηση όπως προβλέπετε. Τότε θα δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πρόοδο προς τις εναλλακτικές λύσεις. Ως προς τις νέες τεχνολογίες, την παραγωγή, έχουμε πετύχει τίποτα, μπορούμε να, να ταχύνουμε την πρόοδο προς το μέλλον και επομένως είναι πολύ σημαντική αυτή η αξιολόγηση. Τελευταίο, θα γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι ότι η θητεία θα ολοκληρωθεί και θα θέλαμε αυτή η πρόταση να εγκριθεί φέτος. Και έτσι θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Αυτό χρειάζεται η αυτοκινοβιομηχανία και οι επενδυτές στην Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε κυρία Βαλιά. Κυρία Ντάλη, ακούσατε ότι είχαν να πούν οι συνάδελφοι. Ναι, ναι, τους ευχαριστώ για τα όσα είπαν. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σας πω κάτι που απασχολούσε και υποστήριζε πάντα το Κοινοβούλιο. Και σε αυτό συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια όσον αφορά τις εκπομπές. Εντάξει, η μεταγέννηση από το NDC e προς το WLTP σημαίνει θα είναι πιο αξιόπιστε τιμέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς αυτή η, ειλικρίνη για τα πραγματικά στοιχεία. Επομένω. θα πρέπει να δούμε το, ότι θα πρέπει να δείχνουμε την ίδια συνέπεια και να επισχύουν το ίδιο για την αυτοκινητοβιομηχανία και με το καινούργιο σύστημα. Όχι, εγώ δεν θέλω να ευνοήσω μια τεχνολογία εις βάρος κάποιας άλλης. Τα είπαμε αυτά και στις συναντήσεις με τους κοιόδες ηγητές. Ε, θέλω να έχουμε πιο καθαρά αυτοκίνητα. Όταν λέμε για αυτοκίνητα μηδενικών ε, και χαμηλών εκπομπών, μιλούμε για 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο και λιγότερο. Μπορεί να αυτό να επιτευχθεί με κάποιο είδους ε, ε, υβριδικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα υβριδικά ε, ηλεκτρικά, ε, με αυτοκίνητα συμπίεσης. Ποιες είναι έχουμε χαμηλές εκπομπές τώρα, να μην είπε στις λεπτομέρειες, αλλά δεν δικαιολογείται το να δίνουμε την εντύπωση ότι εδώ μας απασχόλησε αυτή τη θητεία η απασχόληση μόνο όταν μιλάμε στα ΜΜΕ. Και αυτά που λέμε στην έκθεση για την απασχόληση είναι ευρύτερη εικόνα για το τι επιπτώσεις έχει η προτινόμενη αλλαγή. Τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με αυστηρότερους στόχους θα έχουμε αύξηση στι στις δυνατότητε δυνατότητες και σε αύξηση της απασχόλησης στις 28 χώρες. Και άρα το 40% μείωση του 2030, λέει η Ευρωπαϊκή θα έχουμε 88.000 θέσεις εργασίας. Και έχουμε και άλλες μελέτες του Delft και λέει ότι θα έχουμε 0,04 και ε, αύξηση, ο τέλος πάντων θα δώσει και το Cambridge Econometrics λέει ότι θα υπάρχει, έχουν επιπτώσεις 200.000 μέχρι το 2020 και μετά λέει μέχρι το 2030 θα μπορέσουμε να έχουμε αύξηση με τις 25% ε, επίτευξη του στόχου και αύξηση της παραγωγής τέλο πάντων. Θα χαθούν οι θέσεις εργασίας, θα χαθούν 70.000 εργασίες και 25.000 εργασίες εργασίας για τις μπαταρίες και λένε τα συνδικάτα ότι θα πρέπει να υπάρχει σφαιρική πολιτική και θα πρέπει οι κυβερνήσεις και η Ένωση για φόρτιση, μπαταρίες, ανακύκλωση να κάνουν κατάρτιση και θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι εταιρείε ε, θέσει απασχόλησης. Να συνεχίσουν να συμμορφώνονται και κατά την αλλαγή. Οπότε θα το δούμε αυτά κατά λεπτό όσον αφορά τι τροπολογίε για μια δίκαιη αλλαγή. Ζητήσαμε στοχευμένα προγράμματα για κατάρτιση των εργαζομένων, και να γίνουν όλα αυτά με κοινωνικό διάλογο των κοινωνικών εταίρων. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνο και τέλο πάντων ελπίζω να είναι παραγωγικέ συναντήσει με του συναδέλφου, με του σκιώδε για να καταλήξουμε σε νομοθέτημα τόσο σημαντικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λίζε, παρακαλώ. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά και γι' αυτό θα ήθελα να ξαναπευθύνω την ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Ντάλη προς την Κομισιόν πώς θα λειτουργήσει ε, η προθεσμία του 2025 και την ε, Μίριαμ Ντάλη θέλω να ρωτήσω πώς ε, βλέπετε το θέμα της διαγραφής της παραμέτρου χρηστικότητας που αντιστοιχεί στο βάρος. Ε, δηλαδή, ε, αν ένα όχημα με έξι θέσεις πρέπει να πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις με ένα μικρό όχημα που, όπου βρίσκεται μόνο ένας οδηγός μέσα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, αλλά θα μπορούσατε να τις είχατε θέσει όταν είχατε το λόγο. Δεν πειράζει, θα κάνω μια εξαίρεση. Παρακαλώ, κύριε Μέτσκερ. Ζήτω συγγνώμη κύριε Λίζε. Προσπάθησα να είμαι σύντομος. Γι' αυτό ε, παρέλειψα την ε, ερώτησή σας. Ναι, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ε, η ασφάλεια για τους ε, κατασκευαστές και η μετάβαση από το NLDC στο WLTP. Ε, είχαμε πίνακες αντιστοιχίας. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι οι κατασκευαστές θα μπορούν ήδη τώρα να δουν ε, τι στοιχεία θα βγάλουν τα οχήματά τους. Πρώτον. Δεύτερον, ο κάθε κατασκευαστής μπορεί τα οχήματά του να τα περάσει από τη δοκιμή για να μετρήσει το αποτέλεσμα WLTP και να ε, διαπιστώσει πόσο κοντά βρίσκεται στον πίνακα αντιστοιχίας. Ε, βέβαια, ο τελικός αριθμός ε, θα είναι σχετικός, αλλά το περιθώριο λάθους στον υπολογισμό θα είναι πολύ μικρό. Το δεύτερο θέμα που έχουμε και που ανέφερε η κυρία Ντάλη είναι υπάρχει η δυνατότητα να εξαπατήσει κανείς το σύστημα όπως ε, έγινε στο παρελθόν. Τα δεδομένα WLTP που συλλέγονται στην αρχή αποτελούν την βάση για την μείωση εκπομπών. Εάν λοιπόν ε, υπάρχει δυνατότητα εξαπάτησης ε, της διαδικασίας να προγραμματιστεί δηλαδή το όχημα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να έχει υψηλές εκπομπές στο WLTP, αυτό ε, θα επηρεάσει τη συνέχεια και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πώς αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο παραποίησης των αποτελεσμάτων ουσιαστικά, δηλαδή όπως είδαμε στο πλαίσιο του NLTC. Το Άλλο σημείο είναι ότι θεωρούμε το βάρος απολύτως απαραίτητο. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Λίζε. Δεν μπορεί κανείς ε, να συγκρίνει μεταξύ τους ε, τα οχήματα έτσι απλά. Όσο προχωράμε όμως στα οχήματα μηδενικών εκπομπών, τόσο λιγότερο θα μας ενδιαφέρει το βάρος. θα διαπιστώσετε ότι θα προσθεθούν πολλές δαπανηρές τεχνολογίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν μείωση γρήγορη των μειώσεων και για τα πιο βαριά οχήματα. Ιδιαίτερα αν είναι οχήματα με κυψέλες καυσίμων ή που να κινούνται με μπαταρία. Το βάρος δεν θα ε, σημαίνει τίποτα τελικά. Ε, θα δείτε λοιπόν ότι η καμπύλη αυτή ε, θα καταλήξει σε ευθεία. Δηλαδή το βάρος δεν θα μας ενδιαφέρει τελικά. Αυτή τη στιγμή όμως μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και κύριε Λίζε. Ε, ζητώ συγγνώμη που ε, δεν απάντησα στην ερώτησή σας. Όσα έχουν τα πράγματα σήμερα, οι στόχοι μας δεν αφορούν συγκεκριμένα οχήματα, αφορούν το σύνολο του στόλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε όμως ε, στόχους για όλους τους κατασκευαστές, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πωλήσει ε, ενός έτους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε το βάρος ως δικαιολογία λέγοντας ότι τα μεγάλα οχήματα μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους ανθρώπους. Διότι στο μέλλον θα έχουμε οχήματα με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ακόμα και αν είναι πιο βαριά από άλλα οχήματα. Θα ήθελα πολύ να καταλήξουμε να εξετάσουμε τον συνολικό κύκλο ζωής όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά βέβαια αυτό θα γίνει σιγά σιγά και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ήδη τώρα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, και έτσι ολοκληρώνουμε την συζήτηση. Θα ψηφίσουμε στην ΕΝΒΗ στις 10 Σεπτεμβρίου. Και ε, το θέμα αυτό θα πάει και στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Και το τελευταίο θέμα στην πρωινή μας συνεδρίαση ε, σήμερα το πρωί είναι αντίρρηση ε, που αφορά την ακεταμιπρίδια χρήση σε βιοκτώνα του τύπου προϊόντων 18. Εξετάζουμε πρόταση ψηφίσματος ε, και η συγκήτρια είναι η κυρία Κοντάν. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, παρουσιάζω και πάλι μία αντίρρηση σε σχέση με την έγκριση ενός νεανοκατοειδούς, ενός εντομοκτώνου που ε, ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού των μελισσών στην Ευρώπη. Εδώ πρόκειται για την έγκριση καταμυπρίδης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτώνα προϊόντα τύπου 18 θα ε, χρησιμεύσει για ε, να καταπολεμήσει τα κάρια και τα έντομα που έρχονται ή πετούν και μέσα στα κτίρια αλλά και εξωτερικά στην εξωτερική περίμετρο των κτιρίων. Αυτό το είδος ε, της χρήσης θέτει τα ίδια προβλήματα με την χρήση της ακεταμυπρίδης της καλλιέργειας. Αυτή η ουσία επιτίθεται στο νευρικό σύστημα των μελισσών της που προσανατολίζει και τι σκοτώνει. Θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό των μελισσών, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουμε και να πλαισιώσουμε τη χρήση που γίνεται στο εξωτερικό. Η Κομισιόν μας προτείνει ε, σήμερα να διευρύνουμε τις δυνατότητες χρήσης ε, προϊόντων ε, που ευθύνονται άμεσα για την εξαφάνιση των μελισσών. Ε, θα θυμάστε ότι το Μάρτιο του 2018 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε με βρία πλειοψηφία ένα ψήφισμα για τις ε, προοπτικές και τις προκλήσεις για τη μελισσοκομεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλούσαμε την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση βάσει της επιστημονικής γνωμοδότησης που απαγόρευε τα ανενοικοτοειδή και τα συστημικά εντομοκτώνα να είμαστε λοιπόν συνεπείς. Την στιγμή που θα ψηφίσουμε αυτή την αντίρρηση, η μυπηρίδη δεν διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται για μια ουσία όπου οι επικονιαστές και οι μέλισσε δεν έχουν εκτεθεί ακόμα. Ε, έτσι λοιπόν, ακριβώς ε, ε, σήμερα οι μέλισσες μπορούν να επισκεφθούν ε, τα χωράφια και τις καλλιέργειες και να εκτεθούν ε, σε αυτές τις ουσίες. Ε, η επιστημονική άποψη σε σχέση με τη χρήση της ακτινοπυρίδης είναι ξεκάθαρη. Σε αυτή η ουσία ε, συνεισφέρει πάρα πολύ στην εξαφάνιση των μελισσών στην Ευρώπη. Σήμερα οι μελισσοκόμοι στην Ορμανδία, στη Γαλλία, έκαψαν λόγω της εξαφάνισης ε, των μελισσών τους πάνω από 300 ε, κυψέλες. Έτσι λοιπόν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και σας ζητώ να υποστηρίξετε την αντίρρησή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι παρόντες. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πιέκτα, γιατί ο χρόνος περνάει. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά την ε, Ακετά Μυπρίδη, η Κομισιόν που επέτρεψε τη χρήση αυτού του βιοκτόνου σε θερμοκήπια, ε, έχει γίνει ε, αυτό βάσει της επαρκούς ε, τεκμηρίωσης έχουμε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τους κινδύνους. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι είχε αρνητικέ επιπτώσει στα θερμοκήπια. Όταν όμω μιλάμε για τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ανοιχτού χώρου, υπάρχουν κάποιε εμφιβολίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζει τώρα τις συνέπειες, τα αποτελέσματα των νοικοτινοειδών. Η εκεταμιπρίδη είναι μια τέτοια ουσία που έχει επιπτώσεις στις μέλησεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσισε την απόφασή της για τη χρήση σε θερμοκήπια σε πληροφορίες βάσει των οποίων δεν υπήρχαν κίνδυνοι γνωστοί της ουσίας αυτής για τις μέλισσες. Βέβαια, διαφέρει η κατάσταση αν χρησιμοποιείται το προϊόν σε θερμοκήπιο ή σε ανοιχτούς χώρους. Οι πληροφορίες πάντως ε, δεν είναι πλήρης στην περίπτωση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι οι μελλοντικέ αποφάσεις ε, για την χρήση ή την απαγόρευση αυτή τη ουσία σε ανοιχτού χώρου ε, χρήζει περαιτέρω επιστημονικών ελέγχων καθώς και γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Η την απαγορευση αυτης της ουσιας σε ανοιχτου χωρους χρηζει περαιτερω επιστημονικων ελεγχων καθως αναλυθεί από τα κράτη-μέλη και είναι σχεδόν ομόφωνα τα κράτη-μέλη στην απόφασή τους ε, να επιτρέψουν τη χρήση της ε, και τα μυπρίδης ε, σε κλειστά περιβάλλοντα, σε θερμοκήπια λοιπόν και το υποστηρίζουμε αυτό. Η ομάδα μου, το ECR, καλωσορίζει το γεγονός αυτό και είμαστε επίσης ικανοποιημένοι που μπορούμε να ελέγξουμε τον κίνδυνο στο περιβάλλον ε, και στην υγεία όταν έχουμε χρήση σε κλειστά περιβάλλοντα. Σε τέτοιε συνθήκε θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε και τα μπρίδια, επομένω δεν θα υποστηρίξουμε το αίτημα τη εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάρεντ για την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να αναφερθώ καταρχήν ε, σε κάποια σημεία στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκοντίν στη δήλωσή της ΕΛΑ και στο σχέδιο ψηφίσματος. Καταρχήν δεν είναι ορθό ότι δεν ε, είναι στην αγορά η Εκεταμιπρίδη. Είναι μια υφιστάμενη δραστική ουσία και δυνάμει το κανονισμό περιβιοκτώνων ε, είναι στην αγορά από το 2000 και χρησιμοποιείται. Δεν πρόκειται για νέα εισαγωγή. Το αντίθετο με αυτή την έγκριση, η Κομισιόν περιορίζει τις πιθανές χρήσεις σε σχέση με το τι είναι δυνατό σήμερα, καθώς για τις σημερινές δραστικές ουσίες τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες που έχουν, εάν έχουν. Έτσι λοιπόν, με αυτή την απόφαση έγκριση θα περιορίσουμε τις πιθανές χρήσεις σε σχέση με την κατάσταση σήμερα. Επίσης, δεν είναι σωστό να πούμε ότι αυτό αφορά τη χρήση βιοκτώνων και μπορεί να συγκριθεί με τη χρήση ε, φυτογενομικών προϊόντων. Εδώ εγκρίνουμε την ε, χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όπως ε, τόνισε ο κ. Πίχα. Μιλάμε για την χρήση σε σπίτια και σε περιοχές κοντά σε σπίτια, όχι δηλαδή στους αγρούς ή σε μέρη όπου ε, χρησιμοποιούμε φυτογενομικά προϊόντα. Επίσης, ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων αξιολόγησε τους πιθανούς κινδύνους για τις μέλισσες από τις χρήσεις ε, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αναμένονται πολύ χαμηλοί κίνδυνοι ε, ή σχεδόν καθόλου κίνδυνοι και σίγουρα όχι από τη χρήση σε κλειστού χώρους μέσα στα σπίτια. Έτσι λοιπόν έχει εξολογηθεί πλήρω ο κίνδυνο για τι μέλισσε και θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλό. Στο ψήφισμά τη η κυρία Γκοντίν αναφέρεται και στο εκτιμώντας 12 και ε, ισχυρίζεται ότι η απόφασή μα ε, δεν συνάδει με το πνεύμα τη αιτιολογικής σκέψης. Ούτε αυτό είναι σωστό, γιατί η αιτιολογική σκέψη 12 σχετίζεται με τις ε, ουσίε που υποβάλλουμε δυνάμει των κριτηρίων cut-off, όπω λέγεται, και δεν ισχύει αυτό γιατί είναι κατά μυπρίδη. Συνοψίζοντα η ουσία έχει αξιολογηθεί πλήρω όπω προβλέπεται στον κανονισμό, ο οργανισμό Χημικών έχει εγκρίνει ε, συστήνει την έγκριση και η Κομισιόν αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύσταση αυτή. Έτσι λοιπόν δρούμε ε, πλήρως ε, σεβόμενοι το πνεύμα του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ και να σας ενημερώσω ότι αυτό το σημείο θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα και ίσως τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν, ε, ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.